So, good morning. Ladies Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε στην συνεδρίασή μας. Οι παρόντες είναι ήρωες, δικαιούνται δωρεάν γεύμα μεσημέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με λίγο λεπτή καθυστέρηση. Ναι και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις από ό,τι βλέπω για την ημερήσια διάταξη την εγκρίνουμε. Σημείο 2 ανακοινώσει δεν υπάρχουν ανακοινώσει. Σημείο 3 αν δεν υπάρχουν σχόλια μέχρι το πέρας συνεδρίασης τα πρακτικά της 8ης, 9ης Οκτωβρίου, 6ης Δεκεμβρίου και 28ης Ιανουαρίου θα θεωρηθούν ασυγκεκριμένα. Και περνάμε στο σημείο 4. Δεύτερη εξέταση τη σύσταση προς το Συμβούλιο για τη νέα συνολική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουσβεκιστάν. Και τώρα σας μιλάω ως εισηγητής. Η τρέχουσα συμφωνία ισχύει από το 1999. Οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία ξεκίνησαν στις 23 Νοεμβρίου του 2018. Η Επιτροπή μας πολύ γρήγορα κινήθηκε για να δώσει συστάσεις προς τους διαπραγματευτές. Η πρώτη παρουσίαση έγινε στις 21 Ιανουαρίου και κατατέθηκαν συνολικά 142 τροπολογίες. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνεδρία των συντονιστών στις 6 Φεβρουαρίου και καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε ένα κείμενο που λαμβάνει υπόψη τη συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων των συναδέλφων. Μάλιστα, καταρτήσαμε 19 συμβαστικέ τροπολογίε που αφορούν κυρίω τα ανθρώπινα δικαιώματα, του πολιτικού κρατούμενου, την ελευθερία έκφραση και την καταναγκαστική εργασία. Και από τη στιγμή που θα κληθούμε να δώσουμε τη συγκατάθεσή μα οι συστάσει θα θεωρηθούν ω κριτήρια αξιολόγηση για το κατά πόσο πληρούνται ή όχι οι προποθέσει που θέσαμε από την Ουσμπεκική κυβέρνηση. Αυτά από μένα εν είδη σύντομη εισαγωγή. Θα δώσω το λόγο τώρα στου και ηγητέ, αρχέ γενομένε από τον κύριο Μπράντο Μπενιφέη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την εξαιρετική συνεργασία για τον ε, φάκελο αυτό και γιατί συμπεριλάβατε πολλές από τις ε, τροπολογίες και συμβαστικές προτάσεις μας. Τα τελευταία χρόνια στο Ουσμπεκιστάν χάρη στη νέα πορεία που ανέλαβε ο πρόεδρος Μιτζιλόγεφ ε, δείχνει ότι η συμφωνία αυτή θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο χάρη και στην δική μας συμβολή και που θα ψηφίσουμε σήμερα. Η συμφωνία αυτή δίνει μία περαιτέρω όθηση στην μεταρρυθμιστική προσέγγιση της νέας κυβέρνησης του Ουσμπεκιστάν με αύξηση της εργασίας με τις άλλες χώρες της περιοχής και μεγαλύτερο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Ιδίω σε ό,τι αφορά την κατάργηση της ε, εξαναγκαστικής εργασίας, ένα διαθωτικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, στο ανάντι, όπως και σεβασμό μειονοτήτων, ελευθερία έκφρασης, απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου που επισκέφθηκε την χώρα και μπορώ να βεβαιώσω ότι υπάρχουν όντως βήματα προόδου που έχουν γίνει. Μια, για το τελευταίο θέμα που ανέφερα, τους πολιτικούς κρατουμένους, μπορώ να σας πω ότι με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι πολλοί κρατουμένοι απελευθερώθηκαν. Έχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα στον τομέα αυτό. Θέλω να υπογραμμίσω εξ ονόματος της ομάδας μου ότι θεωρούμε αναγκαίο να συνεχίσουμε να δεσμευόμαστε υπέρ της απελευθέρωσης και άλλων πολιτικών κρατουμένων. Ευχαριστώ και καλή δουλειά. Thank you, Mr. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπενιφέη. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Τσάρλς Στάνοκ. Δυστυχώς δεν ακούγεται το μικρόφωνο του κύριου Τάνοκ. Ε, δεν έλαβα την ημερήσια διάταξη γιατί μιλάμε για το Ουσμπεκιστάν. Συμφωνώ απόλυτα με τον προλαλήσαντα, τον κύριο Μπενιφέη. Ε, εδώ και χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση στη χώρα αυτή και έχουμε διανύσει μεγάλο δρόμο από τότε που η προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Καρίμοφ κατηγορήθηκε για φρικαλαιότητες, ε, ακόμη και για ε, το ότι έκαψε ζωντανό έναν κρατούμενο Επίσης υπήρχαν κατάφορε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασία παιδιών κατά τη διάρκεια των, της, Οπότε ε, νομίζω ότι τώρα μετά την πρόοδο που έχει σημειωθεί είναι σημαντικό να συνάψουμε τη νέα συνολική συμφωνία και να συσφίξουμε τις σχέσεις μας ε, με τη χώρα αυτή που είναι η πιο πολυπληθής ε, και ηγετική χώρα στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Γι' αυτό και στείλω την έκθεση και μετά από αυτά που άκουσα και από τον εισηγητή μπορώ να σας διαβεβαιώσω για την υποστήριξη της ομάδας των συντηρητικών μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ, Τσάρλς. Ο Χέλμοντ Σόλς, μια και απουσιάζει ο συντονιστής, ο σκιώδης της Άλντε. Ευχαριστώ, κύριε Σιγητά. σε ό,τι αφορά αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, που μας έχετε παρουσιάσει. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με πολλά. Θεωρώ ότι οι εξελίξεις στο Ζουμπεκιστάν ε, έχουν καταγραφεί με πιστό τρόπο Σίγουρα υπάρχουν πολλές προκλήσεις ε, για την ε, περαιτέρω ε, διαμόρφωση των σχέσεων των δύο πλευρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουσμπικιστάν. Βέβαια, πολλές είναι υποχρεώσεις της ίδιας της χώρας. Έχουμε καταθέσει αρκετές τροπολογίες όπου αναφερόμαστε στην ακόμη μη ικανοποιητική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Έχουμε και την κακή κοινωνική και περιβαλλοντική κατάσταση που επίσης ε, έχουμε αναφέρει στις τροπολογίες μας και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε πιθανή αναβάθμιση των σχέσεων ε, και στην περαιτέρω εξέλιξη και πρόθεση της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης και Συνεργασίας, πώς θα το δούμε, πώς ε, θα επηρεάσουμε αυτές τις αναπτυξιακές διαδικασίες. Σίγουρα υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο έκθεσης και στο βαθμό που συμπεριλαμβάνονται, εμείς θα υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ τον Χέλμουντ Σόλτς, έλεγε ο πρόεδρο. Ο Μιχαήλ Γκάλερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο ένα ειδικό συγκεκριμένο σημείο θέλω να αναφέρω σε ό,τι αφορά τις συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες. 13 νομίζω υπάρχει κάτι που δεν έγινε κατανοητό. Έχει ληφθεί υπόψη επί της ουσίας η δική μου τροπολογία, αλλά αν κανείς δει συγκεκριμένα το κείμενο λέει ότι ζητείται η συμβόλη των εθνών εταίρων ώστε η δημοκρατία του Ουσβεκιστάν να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις ε, της καταστροφής ε, στην λίμνη Αράλη και τα είδαμε είναι μια αυτόνομη ε, δημοκρατία αυτή η περιοχή εκεί ανήκει και πρέπει οι αρμόδιοι να έχουν ε, την ε, υποστήριξη στο συγκεκριμένο θέμα. Εντάξει, σίγουρα το Ουσμπεκιστάν στο σύνολό του, αλλά με τη δική μας την τροπολογία εννοούσαμε συγκεκριμένα αυτή την αυτόνομη δημοκρατία Καλπαστάν. Άρα πρέπει να διαγραφεί. Κάρα Καλπακστάνη κάπως έτσι γιατί είναι δύσκολο το προφέρω στη θέση του ε, Ουσμπεκιστάν. Μάλλον παρόραμα ήταν ε, όταν ε, μεταφέρθηκε η ε, δική μου διατύπωση στη συμβαστική τροπολογία. Επαναλαμβάνω, 13 συμβιβαστική. Are you aware of this 13? Την έχετε υπόψη αυτή την συμβιβαστική 13 Λέει ο πρόεδρος. Καλύπτει, λέει ο κ. Γκάλερ, την τροπολογία 88 που είχα καταθέσει εγώ συγκεκριμένα. Το θέμα είναι η διατύπωση. Δεν λέγεται Καρακαλπαστάν, αλλά Ουσμπεκιστάν. Ο στόχος μου ακριβώς ήταν να είμαι συγκεκριμένος και να αναφερθώ στη συγκεκριμένη αυτή ε, αυτόνομη δημοκρατία, όπως είπα. Years Ξέρετε, πριν πάρα πολλά χρόνια είχα μιλήσει για την απερίμωση της Λίνης Αλ και το λαό αυτής της αυτόνομης δημοκρατίας ε, και πραγματικά ε, το πρόβλημα ε, δεν καταλαβαίνω κατά πόσο μπορεί μόνο από το Ουσμπεκιστάν, αλλά επειδή έχει σύνορα και με το Καζακστάν αυτή η περιοχή, ίσως η Κεντρική Ασία συνολικά θα έπρεπε να κάνει κάτι. Ναι, απλά λέει ο κύριος Γκάλερ, το θέμα είναι το Ουσμπεκιστάν, εξού και το ανέφερα σε αυτή την έκθεση. Από πλευρά Ουσμπεκιστάν δηλαδή, εκεί ε, πρέπει να αναστήσουμε το βασικό μας ε, συνομιλητή για την αντιμετώπιση των συνεπειών αλλά ναι, συμφωνώ επί της ουσίας ότι το θέμα αυτό καθεαυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και σε περιφερειακό επίπεδο, επίπεδο Κεντρικής Ασίας. to... Ευχαριστώ. Οπότε, αν θέλετε να αφαιρέσουμε το Ουσμπεκιστάν και να προσθέσουμε το Καρακαλπακστάν στη Συμβαστική Τροπολογία 13, μπορούμε να το κάνουμε αμέσω ή θα πρέπει να συντάξουμε μια προφορική τροπολογία στη Συμβαστική αυτή το 13. Νομίζω ότι έγινε απλώς λάθος ε, στην ε, μεταγραφή και την κάλυψη της δικής μου τροπολογίας 88 από την ε, συμβαστική τροπολογία. Έγινε λάθος μεταφορά. Κύριε Μπενιθέ, κύριε Σόλ, συμφωνείτε? Και να πούμε ιδίω και μετά να προσθέσουμε το όνομα αυτής της δημοκρατίας του Καρακαλπακστάν. Ουσμπεκιστάν και κυρίως ε, η δημοκρατία του Καρα... Καλπακστάν. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Άλλος κανείς παρακαλώ. Όχι, οπότε θα ακούσουμε τον κύριο Γεροσέβιτς. Είναι παρόν από την, Ευρω... από την ΕΕ. Σμίτελ. Παρακαλώ. Είμαι αρμόδιος για το Ουσμπεκιστάν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην ΑΕΔ. Σας ευχαριστώ που ζητήσατε και τη δική μας γνώμη για αυτή την ε, έκθεση που είναι πολύ επίκαιρη. Πριν από 10 μέρες είχαμε στην Τασκέδη ένα γύρο διαπραγματεύσεων, πήγαν πολύ καλά και οι Ουσμπέκη, η Ουσμπεκική πλευρά ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη. Γι' αυτό και καταφέραμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο. Διεκπερώσαμε πολλά ε, σημεία και σας ε, ενημερώσαμε για τους στόχους και την πορεία των διαπραγματεύσεων, κύριε Πρόεδρε. Εν πάση περιπτώσει, θα κρατάμε ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων και δημονούμε να λάβουμε την οριστική ε, μορφή της έκθεσης. Χαίρομαι που στηρίζετε τις μεταρρυθμίσεις του Ουσμπεκιστάν και τη νέα συνολική συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία, που είναι ένα μέσο για τη στήριξη αυτών των, διαπραγματε... των ε, μεταρρυθμίσεων. Είναι πολύ επικοδομητική η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σχέση με το Ουσμπεκιστάν και την εκτιμούμε ιδιαίτερω. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλον κανέναν. Η ψηφοφορία θα γίνει το απόγευμα, όπως ξέρετε, για το θέμα αυτό και θα ξεκινήσουμε στις τρεις τις ψηφοφορίες. Και μάλιστα στην Ολομέλεια ε, έχει προγραμματίσει το θέμα για τη δεύτερη Ολομέλεια του Μαρτίου. Σημείο 5 τώρα. Εξέταση του σχεδίου συστάσεων προς το Συμβούλιο, ε, την Επιτροπή και την Επατή Εκπρόσωπο για το, τη Συμφωνία Θεσμικού Πλαισίου με την Ελβετία. Μάλιστα, ήδη στις 23 Νοεμβρίου έγινε, ε, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με ένα κοινό κείμενο μετά από τετραετή διαπραγμάτευση. Τελικά η Ελβετία αποφάσισε να ξεκινήσει δημόσιες διαπραγματεύσει 7 Δεκεμβρίου που συνεχίζονται. Σίγουρα η Ελβετία είναι από του ε, στενότερου εξωτερικού μεσεντέρου. 1,4 εκατομμύρια Ευρωπαίων υπηκόων διαβίουν στην, Ευρωπαϊ... στην Ελβετία και 450.000 Ελβετοί υπήκοοι διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελβετία είναι μέρο τη ε, ΖΕΣ αλλά όχι και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οι τρέχουσες διμερείς μας σχέσεις στηρίζονται σε ένα πλέγμα 20 κύριων και 100 δευτερευουσών συμφωνιών και μάλιστα με το, με το νέο θεσμικό πλαίσιο θα αποκαταστήσουμε μια μεγαλύτερη συνοχή ε, στη σχέση μας ε, με την Ελβετία και τη συμμετοχή της στην εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι συνδεδεμένη επιτροπή ε, και με βάση το άρθρο 54 θα πρέπει να εγκριθούν οι τροπολογίες και επίση η Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτή έχει εκδώσει γνωμοδότηση. Ο κύριος Φροντζουλίκα, ο εισηγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Όπως αναφέρθηκε, οι δύο πλευρές είναι στενή εταίροι, οικονομική και πολιτική και καλύπτονται και το εμπόριο των αγαθών και υπηρεσιών και τις άμεσες επενδύσεις. Η συνεργασία μας όμως ξεπερνά την οικονομική διάσταση. Η Ελβετία έχει στενούς πολιτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με την Ένωση και τα κρατημέλη της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελβετία ήταν υποψήφια για μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διέκοψε τη διαδικασία αυτή το 2016. Ωστόσο, οι αμοιβαία θετικές σχέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν κοινή ευθύνη για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των σχέσεών μας. Γι' αυτό ήθελα η έκθεση να είναι ισορροπημένη, παρέχοντας ε, μια ισορροπημένη προσέγγιση για τις απόψεις όλων και ε, συμβάλλοντας με σωστές προτάσεις στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την είπα εκπρόσωπο. Η Ελβετία είναι στενός εταίρος, θέλουμε να γίνει στενότερο στο μέλλον. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελβετίας και της Επιτροπής για το, τη Συμφωνία Θεσμικού Πλαισίου ξεκίνησαν το 2014 και ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2018. Δυστυχώς, στις 7 Δεκεμβρίου του 2018 το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας αποφάσισε ούτε να δεχθεί ούτε να απορρίψει την ε, συμφωνία αλλά ζήτησε να γίνει μια δημόσια διαβούλευση για το επόμενο εξάμεινο. Οι διμερείς σχέσεις των δύο πλευρών είναι σημαντικές μια και υπάρχουν πάνω από 120 διμερείς συμφωνίες που ισχύουν αυτή τη στιγμή και συμβάλλουν ε, σημαντικά στην ευημερία όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Γι' αυτό είναι προς το συμφέρον και των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του λαού της Ελβετίας να εξασφαλιστούν στο μέλλον οι διμερείς αυτές τις συμφωνίες μέσω ενός θεσμικού πλαισίου. Γιατί κυρίε και κύριοι συνάδελφοι υπάρχουν κάποιες συμφωνίες οι οποίες ανατρέχουν το, στο 1974 που είναι πλέον ε, και πρέπει να ενημερωθούν. Μέχρι τώρα το πλαίσιο συμφωνίας που διαπραγματεύεται ε, δημιούργησε κάποιες διαφορές, ιδίως στον τομέα των οδηγιών για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και της προστασίας των ε, μισθών, ε, ιδίως με την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Η διαφορά απόψεων εμφανίστηκε στο πώς αυτό αντικατοπτρίζεται στην έκθεση. Υπήρξαν πολλές εξωτε... πολλά εξωτερικά αιτήματα από διάφορους οργανισμούς και φορείς να υιοθετηθεί στην έκθεση μία πιο μετρημένη προσέγγιση στα μονομερή μέτρα που υιοθέτησαν οι Ελβετοί για την προστασία των Ελβετών εργαζομένων από το κοινωνικό ντάμπιγκ και να φύγουν οι αναφορές που έλεγαν ότι αυτές οι διατυπώσεις ήταν, ε, αυτές οι διατάξεις ήταν ε, διακριτικού χαρακτήρα. Ως υπήρξαν 76 τροπολογίες, κάποιες από αυτές δικές μου, που καλύπτουν όλες τις διαφορές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους Κιώδης για τη συνεργασία τους. Κάναμε δύο γύρους ε, συνεδριάσεων των σκιωδών εισηγητών. Ε, παραμένουν βέβαια κάποιες, ε, συμφωνίες, κάποιες διαφωνίες στην αναφορά στο συμβιβαστικό 4, όπου κάποιοι θεωρούν ότι η αναφορά στις μονομερείς αυτές, ε, στα μονομερή αυτά μέτρα δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση. Είναι γεγονός ότι τα συνοδευτικά μέτρα είναι μονομερή. Υιοθετήθηκαν δηλαδή μόνο από την ε, Ελβετία. Δεν ευθυγραμμίζονται με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς και δεν είναι συμβατή, συμβατά με την ελεύθερη κυκλοφορία. Ιδίω σε ό,τι αφορά τους ε, εργαζόμενους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσπασμένους και ελεύθερους, είναι, είναι φανερό ότι δεν είναι ε, αναλογικά. Η... Τα μέτρα αυτά δεν θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και ο κανόνας θα έπρεπε να ισχύει για όλους με όμοιο τρόπο στην εσωτερική αγορά. Η άλλη άποψη οδηγεί στην αποχώρηση από την εσωτερική αγορά. Το στόχο των συνοδευτικών μέτρων είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού dumping στον τομέα των υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ωστόσο με μέτρα που μπορούν να στηρίζονται στους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας. Δείξατε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πολύ έφεση δουλειά και το κείμενο της συμφωνίας δίνει έμφαση σε μέτρα που είναι συναφή με τα συνοδευτικά ούτω ώστε το, το, το, παρόν κείμενο δεν καλύπτει την, τις μελλοντικές σχέσεις. Η, Ελβετία συνεχίζει να βρίσκεται στη διαδικασία διαβουλεύσεων, αλλά τα υφιστάμενα μέτρα ισχύουν. Τελειώνοντας, συνάδελφοι, θέλω να υπογραμμίσω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου χθε για την Ελβετία. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και παραθέτω λένε το Συμβούλιο λυπάται ιδιαίτερα διότι το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας δεν υποστήριξε την έκβαση των διαπραγματεύσεων του, της 7ης Δεκεμβρίου και ζητά από το Συμβούλιο να ξεκινήσει την ε, διαπραγμάτευση του κειμένου υποβάλλοντας προς έγκριση το κείμενο αυτό στο ομοσπονδιακό, στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση των εμπλεκομένων φορέων την άνοιξη του 19. Συμπερασματικά το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ανησυχία της για την ασυνεπή εφαρμογή κάποιων συμφωνιών και την εφαρμογή από την Ελβετία ε, μεταγενέστερων μέτρων που είναι ασύμβατα με τις συμφωνίες, ιδίως την ε, συμφωνία για αμοιβαία συνδρομή. Στο, συμβούλιο αυτό το, στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο ζητά από την Ελβετία να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ιδίως στο θέμα των αποσπασμένων εργαζομένων και στους παρέχοντες υπηρεσία στο έδαφος της με βάση τις ευρωπαϊκές αρχές της, της αναλογικότητας και της μη διάκρισης. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε και τώρα θα δώσω το λόγο στους κοιόδης συζητητές. Τα κυρία Ζέλανα Ζόφκο. Ευχαριστώ. Ε, με ιδιαίτερη χαρά ανέλαβα να παρακολουθήσω και οδησυγήτρια αυτή την έκθεση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φροζούλικα για την προσέγγιση που είχε στις ε, διαπραγματεύσει για τις συμβαστικέ τροπολογίες. Ευχαριστώ και τους λοιπού και οδησηγητέ. Είχαμε πραγματικά εξαιρετική συνεργασία. Το νέο θεσμικό πλαίσιο και σχετική συμφωνία που ε, ξεκινήσαμε να διαπραγματευόμαστε το 2014 μέχρι πέρυσι είναι ευπρόσδεκτη. Δυστυχώ ακόμη η Ελβετία δεν κύρωσε το κείμενο που περιλαμβάνει και ένα δημοψήφισμα. Ενθαρρύνουμε λοιπόν με την έκθεση το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετία να εγκρίνει το κείμενο που είναι το αποτέλεσμα τη διαπραγματεύση. Δεν θέλω να σταθώ σε ένα σημείο που είναι ιδιαίτερα προσφυλέ για μένα. Ζητούμε από την Ελβετία να μειώσει την περίοδο ε, μεταφορά ε, εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων για τους Κροάτες εργαζόμενους. Πρόσφατα αποφασίστηκε η παράταξη της αρχικής ε, διετίας ε, και παρόλο που έχει σταθεροποιηθεί η ροή από την Κροατία. Επίσης και η θέση του Συμβουλίου λυπάται για την θέση αυτή της Ελβετίας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι τα γνωστά ως συνοδευτικά μέτρα. Το 2004 τα εισήγαγε η Ελβετία για να προστατεύσει τις επιχειρήσεις από το δάμι και τον αθέμητο ανταγωνισμό. Βέβαια δεν συνάδει με την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και ανθρώπων. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται δήλωση 8 ημέρες προηγουμένω και να πληρώνουν ειδικό τέλος οι εταιρείε. Και μάλιστα συχνά γίνεται έλεγχο ε, των ε, ε, ευρωπαϊκών εταιριών σε αντίθεση με 3% μόνο των ελβετικών εταιριών παρά το ίδιο επίπεδο παραβιάσεων. Είναι σαφή και κατάφορη αυτή η δυσανάλογη και δυσμενή μεταχείριση βάρο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Επίση, τι γίνεται με του Ευρωπαίου υπηκόου που μένουν στι παραμεθόρειε περιοχέ. Γι' αυτού ακριβώ διαπραγματευτήκαμε αυτή τη νέα συμφωνία πλαίσιο. Λυπάμαι για τη θέση τη Ελβετία όπω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σίγουρα είναι συνοπτική και άρτια έκθεση που δείχνει ότι θέλουμε ε, μόνιμες ε, και καλές σχέσεις με την Ελβετία και είμαστε υπέρ της έγκρισης της ε, συμφωνίας που πιστεύω ότι θα ωφελήσει και τα δύο συμβαλωμένα μέρη και κυρίως τους πολίτες τους. Ευχαριστώ. Κύριε Στάνο, και επόμενος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Φουντζουλίτσα για την εξαιρετική του έκθεση χρησιμοποίησε τις λέξεις ε, στενός εταίρος της Ένωσης για την Ελβετία. Δεν ξέρω αν θα ήθελε η ουδέτερη Ελβετία να αναφέρεται αυτή η διατύπωση, γιατί δεν συμμετέχει σε στρατιωτικέ εταιρικέ σχέσει ε, ε, στην πολιτική ασφάλεια. Είναι σίγουρα ένα στενός εταίρος σε πολλά άλλα μέτωπα. Τέσσερις ε, χώρες, ε, μεταξύ των οποίων και τα Φερό, έχουν συνάψει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο ε, πριν από τον Brexit και η Ελβετία βέβαια και πολλοί θεωρούσαν ότι το ελβετικό μοντέλο ήταν αυτό που θα είχε εγκριθεί από τη Βρετανία. Όταν όμως ανακάλυψαν ότι περιλαμβάνει ελευθερία προσώπων δεν τους άρεσε και πολύ, ελευθερία διακίνησης δηλαδή. Και στην ΕΖΕΣ έγινε, ενώ ήταν μέλος της ΕΖΕΣ, η Ελβετία έκανε αυτό το λαϊκό δημοψήφισμα και δεν ε, ψήφισαν οι Ελβετοί να γίνει μέλος ε, της Ένωσης. Ε, υπάρχει όλες αυτές οι εμπορικές και άλλες 20 και άλλες συμφωνίες και δεν υπάρχουν μόνιμα δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν διάφορες διαφορές και δεν ξέρω κατά πόσο ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε και μιλάω βέβαια πάλι για τη Βρετανία να ακολουθηθεί στη μετά την Brexit εποχή. Εγώ θα στηρίξω τις συμβαστικέ και ελπίζω να περάσει με μεγάλη πλειοψηφία αυτή η έκθεση. Πιστεύω ότι αυτό είναι δεδομένο. Ευχαριστώ. you, Σε ευχαριστώ. Ο πρόεδρος δεν υπάρχει άλλος σκιώδης που να ζητά το λόγο τουλάχιστον. Επομένως, Περνώ στους λοιπούς ομιλητές. Ο κύριος Ντόρμαν είναι εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο της ε, αντιπροσωπείας και ασχολούμαστε με τα θέματα της ε, Ελβετίας. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης και τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες που νομίζω ότι υποστηρίζονται από την ευρεία πλειοψηφία της Επιτροπής μας. Ε, οι διαπραγματεύσει μεταξύ Ελβετίας ε, και Ελβετίας και Ευρωπαϊκής πήγαν πολύ καλά και οι διαπραγματές ε, των δύο πλευρών λειτουργήσαν καλά. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ καλό κείμενο μπροστά μας, ιδίως το άρθρο 16 με ικανοποιεί αυτής της συμφωνίας για την κοινή Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ελπίζω σύντομα να αναβαθμιστεί το EPM που είναι στη δική μας την αντιπροσωπεία. Έχουμε όμως και εκλογές και στην Ένωση και στην Ελβετία. Είναι κάπως πολύπλοκα λοιπόν τα πράγματα. Το EFA θα βελτιώσει περαιτέρω τις οικονομικές σχέσεις που έχουν ωφέλη να προσφέρουν και στις δύο πλευρές. Και είναι και σημαντικός παράγοντας αυτή η συμφωνία πλαίσιο και σε Συμφωνία για την Πρόσφαση Αγορές. Εκφράζονται διάφορες απόψεις. Πρόσφατα επισκέφθηκα την Ελβετία και το διαπίστωσα. Ο επικεφαλής της Ελβετικής Αντιπροσωπείας, Hans Peter Bockmann, είχε μία συνάντηση μαζί μου και είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση και στο Ελβετικό Κοινοβούλιο πήγε πολύ καλή συζήτηση, αλλά έδειξε ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες στη χώρα. Ε, βέβαια, αντίστοιχες ανησυχίες υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ένωσης. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Ντόρμαν. Και θα δώσω το λόγο στους πόμους για Σουίτσα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδρες εισηγητές για το κείμενο αυτό. Μία τροπολογία θα ήθελα να σχολιάσω όλους ιδιαιτέρως ε, την υπαριθμό 45 και ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί κατενόησε το λόγο τον οποίο συγκαταθέτω με τον συνάδελφο Ράντος από την Κροατία αυτή την τροπολογία. Η τροπολογία αυτή λέει, εκφράζει τη λύπτη για το γεγονό ότι η Ελβετία αποφάσισε σε 7 Δεκεμβρίου 2018 να παρατείνει τα μεταβατικά μέτρα για του Κροάτε εργαζομένου πέραν τη αρχική περίοδου των δύο ετών. Και καλή κατά συνέπεια την Ελβετία να εξετάσει το ενδεχόμενο συντόμευση τη περίοδου εφαρμογή των ελόγων μεταβατικών μέτρων, λαμβάνοντα υπόψη τα ωφέλη τη ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετία. Περιλαμβάνει τι συμβαστικέ τροπολογίε. λόγω το Σα ευχαριστώ. Όμως, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι η πρόταση αυτή στο αρχικό της ΚΙΜ περιλαμβάνεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής και Ελβετίας και εγκρίθηκε χθε στη συνεδρία του Συμβουλίου. Αυτό είναι πολύ καλή εξέλιξη και θα υπογραμμίσω. Είναι κάτι σημαντικό για την Κροατία και τους Κροάτες εργαζομένους. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Πίτσουλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά τον εισηγητή μας, τον κύριο Φρουντσουλίκα, για τις ε, πολύ θετικές συμβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα να εκφράσω εγώ την λύπη μου για την ε, παράταση της προθεσμίας των μεταβατικών μέτρων για τους Κροάτες εργαζόμενους και για την πρόσβασή του στην ελβετική αγορά εργασίας και μετά την εκπνοή της πρώτης φάσης και την υιοθέτηση του τρίτου πρωτοκόλου. Κάτι τέτοιο παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας. Και μάλιστα ε, την 1η Ιανουαρίου του 2017 πρότεινε παράταση κατά άλλα τρία έτη. Ε, και το Συμβούλιο εξέφρασε την ε, δυσαρέσκειά του με την απόφαση αυτή. Και μάλιστα η συμβαστική μας τροπολογία παρόλο που είναι κάπως πιο ήπιες διατύπωσης, ε, καλύπτει αυτό το θέμα. Ε, οι Κροάτες εργαζόμενοι έχουν μια καλή ενσωμάτωση στην ελβετική αγορά και η ανεργία τους είναι χαμηλότερη από το κοινοτικό μεσόωρο. Ε, κάτι που επιβεβαιώνει την πολύ καλή ενσωμάτωση τους στην κοινωνική τους ένταξη και την ένταξη στην, εργασιακή τους, στην αγορά εργασίας της Ελβετίας. Άλλωστε είναι μικρός ο αριθμός των κρατών εργαζομένων, 0,02% σε σχέση με το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό. Φαντάζομαι ότι κάποιοι συνάδελφοι λαμβάνουν από τα συνδικά τους άλλα μηνύματα και έχει πολιτικοποιηθεί ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα της προσαρμογής. Αλλά εδώ δεν μιλούμε μόνο για ποσοστά και απόλυτους αριθμούς. Εδώ μιλούμε για ίση μεταχείριση όλων των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης μιλούμε για την αμοιβαιότητα των σχέσεων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες με τις οποίες έχει συμφωνίες και στενέ σχέσει Γι' αυτό ζητώ από την Ελβετία να δείξει κατανόηση και φυσικά τους συναδέλφου να δείξουν κατανόηση και ευχαριστώ και πάλι για την ε, έκθεση τον κύριο Φρουντζουλικά. Ε, Ευχαριστούμε. Κύριε Ζόφκο ζήτησε να προσθέσει κάτι. Και εγώ θέλω να συμφωνήσω με τον συνάδελφο από την Κροασία και να τον διαβεβαιώσω ότι μαζί με τους άλλους και όλους εισηγητές φροντίσαμε να συμπεριληφθεί πλήρως η τροπολογία για τους ε, αποσπασμένους εργαζομένους στη συμβαστική πρόταση και υποστηρίζεται όλες, από όλες τις ομάδες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτς έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. σε ό,τι αφορά τη θέση του εισηγητού και των σκιωδών εισηγητών, πολλά είναι αυτά τα οποία πηγαίνουν προ σωστή κατεύθυνση. Μιλάμε για μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία, οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών και το πώς θα προχωρήσουν και πώς πρέπει να εξελιχθούν περαιτέρω. Υπάρχει όμως αυτή η συμφωνία και η διάσταση ε, του Brexit και το πώς θα διαμορφωθεί μελλοντική σχέση και αν υπάρχουν αναλογίες σε ό,τι αφορά τους μισθούς, σε ό,τι αφορά την ελευθερία μετακίνησης, ε, ε, των εργαζομένων, ελεύθερη κυκλοφορία, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη και η παροχή υπηρεσιών και πρέπει να ακούσουμε την άποψη των ε, ελβετικών εργαζομένων και των ελβετικών συνδικάτων. Υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια πολύ αυστηροί κανόνες ε, εγγύησης και το τι μέτρα πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στην Ελβετία. Όλα αυτά μπορεί να αποδυναμωθούν, είναι ένα κίνδυνο. και υπάρχουν διάφορα ε, απαράδεκτα κατά την άποψή μα ε, στοιχεία στην έκθεση γιατί δεν πηγαίνουν σωστή κατεύθυνση. Παραδείγματο χάρη σε μια ε, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου υπάρχει ένα κεφάλαιο αηφορία με πολύ συγκεκριμένου όρους και προϋποθέσεις κατά την άποψή μας ε, ε, θα πρέπει να περιλαμβάνονται και μέτρα εφαρμογής στις ε, διατάξεις αυτής της συμφωνίας, εκτελεστικά μέτρα. Και στο τρίτο τμήμα για τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή δεν υπάρχει ακόμη κάποια απόφαση τι θα γίνει με τις άλλες ε, ομάδες, ε, τις εγχώριες, ε. τι θα γίνει με τη σχέση εργαζοδοτών εργαζομένων και των υπηκών Ελβετίας και των αλλοδαπών υπηκών που διαμένουν εκεί. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα επεξεργαστούν οι δύο πλευρές έτσι περαιτέρω. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν το λόγο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, ΕΙΕΔ. Ο κύριος Μάρτιν Σκύλ εκπροσωπεί την, Επιτροπή, ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Μάρτιν, πώς λέγεσαι τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την σύστασή του. Η Συμφωνία Θεσμικού Πλαισίου θα είναι αμοιβαία θετική παρέχοντας ασφάλεια δικαίου και ενιαίους κανόνες για πολίτες και επιχειρήσεις ε, στην εσωτερική αγορά. Περιλαμβάνει ε, το, τα βασικά κομμάτια του κεκτημένου και επιτρέπει την, ε, το προδικαστικό ερώτημα προς το Δικαστήριο της Ένωσης. Ταυτόχρονα θα βοηθήσει να λυθούν πολλά εκρεμή προβλήματα. Τώρα, για τα συνοδευτικά μέτρα. Η Ένωση και η Ελβετία έχουν τους ίδιους στόχους. Προστασία υψηλού επίπεδου εργασιακά πρότυπα και μισθούς. Η Ένωση παρέχει τρόπους για να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και την προστασία της αγοράς από μισθολογικό ντάμπινγκ και αθέμητες πρακτικές. Πιστεύουμε ότι τα υφιστάμενα μέτρα όπως τα έχει θεσπίσει η Ελβετία, είναι και διακριτικά και δυσανάλογα, περιορίζοντας την ελεύθερη παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των, των πολιτών εις βάρος των πελατών στην Ελβετία, που έχουν ε, λιγότερες δυνατότητες να αντιμετωπίσουν τις σημερινές υψηλές τιμές. Πετύχαμε ένα καλό συμβαστικό κείμενο στις διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό, καλύπτοντας τις εκκρεμείς ακόμα ανησυχίες των Ελβετών, σεβόμενοι ταυτόχρονα την αναθεωρημένη, την οδηγία 75 του 18 για την απόσπαση των εργαζομένων. Προτείναμε μια σειρά προσαρμογών λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικέ συνθήκες της αγοράς εργασίας της Ελβετίας για την παροχή υπηρεσιών από Ευρωπαίους ε, παρόχους, δεχόμενοι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων να συνεχίσουμε τις απαιτήσει προκοινοποίησης έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες για, για υποκαταστήματα και εξέταση της ανάλυσης με ανάλυση κινδύνου. Εξετάσαμε ταυτόχρονα την παροχή εγγυήσεων πριν την παροχή των υπηρεσιών στην ε, περίπτωση που κάποιοι πάροχοι υπηρεσιών δεν τηρούν τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις. Επίσης, ελέγχους για την, αντιπα... για την μετώπιση της ε, ε, της ε, ταυτόχρονα, δεν αγνοούμε τη σημασία της οδηγίας για την, την, ευρωπαϊκή ηθαγένεια στα πλαίσια της απόσπασης εργαζομένων και, στο, και εδώ θεωρούμε ότι μπορούν να υπάρξουν προσαρμογές όπως αν ε, αναγνωρίστηκαν για χώρες ε, εόχεζες που δεν υποχρεώνουν τις χώρες αυτές να υιοθετήσουν τη, τον ορισμό της ηθαγένειας της Ένωσης στην εθνική του νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ναχτά. Κλείνοντας, ο κύριος Φουντζούλικα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και συναδέλφους εκ νέου. Έκανα ό,τι μπορώ για να εντάξω στις συμβαστικές τοπολογίες όλες τις θέσεις των συναδέλφων. Ε, συμφωνείτε νομίζω ότι είναι μια ισορροπημένη έκθεση που αποσκοπεί στο να προστατεύσει τα συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης και των κρατών της Ένωσης. Αναφέρατε, αναφέρθηκε και το είδατε ότι η Ευρωπαϊκή, ε, είμαστε λίγο πιο ε, επικριτικοί από ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θεωρούμε ότι κάποια μέτρα είναι διακριτικά, αφήνοντας ε, χώρο για περαιτέρω αντιμετώπιση και τονίζουμε την λύπη μας για το ότι η κυβέρνηση της στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δεν υιοθέτησε το Δεκέμβριο τη συμφωνία. Δυστυχώ, διαβάζοντα τον ελβετικό τύπο έχω την εντύπωση ότι δεν θα υποστηρίξουν τη συμφωνία αυτή. Σα το λέω έτσι προκατατικά. Τέλο πάντων, εμεί τη δουλειά μα την κάναμε προστατεύοντα τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΑΦΕΤ ε, θα γίνει σήμερα το απόγευμα και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο, στο επόμενο σημείο το 6 αλλά σε αντίθεση με άλλες φορές ε, διεκπαιρώνουμε πολύ γρήγορα τα σημεία και νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ε, και μου λένε ότι δεν είναι παρόντες ακόμη οι ομιλητές μας ε, για το σημείο 6, γι' αυτό μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο 7 προς το παρόν. Ο κύριος Χαουρέγγι μου είπαν ότι έρχεται. Πού είναι ακριβώς όμως, σε ποιο σημείο βρίσκεται. Γνωρίζει κανείς. Can somebody call him? Μπορεί κανείς να το τηλεφωνήσει παρακαλώ. Εμένα είναι τα Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάνουμε, όπως είπα και πριν, στο σημείο 7. Θα μας ενημερώσει ο κύριος Χαουρέγγι για τα όσα συνέβησαν στην αποστολή. Ήταν επικεφαλής ο κύριος Χαουρέγγι της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ικαράγουα. Επτά μέλη ήταν η αντιπροσωπεία και μάλιστα στόχος ήταν να γίνει μια εκτίμηση της κατάστασης επί τόπου και να στηρίξουμε τον πολιτικό διάλογο μετά την κρίση που ανέκυψε και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χωρίς άλλη χρονοτριβή θα δώσω το λόγο στον κύριο Χαουρέγγι, ευχαριστώντας τον που έσπευσε να έρθει και νωρίτερα από ό,τι προγραμματιζόταν το δικό του σημείο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όντως πρέπει να σας ενημερώσω ότι η αποστολή στην Ικαράγουα έγινε 23 με 26 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους. Η αποστολή ήταν πολύ σημαντική από πολιτική άποψη, αλλά και πολύ συγκινητική από προσωπική άποψη. Γιατί καταφέραμε να διαπιστώσουμε η μας τι συμβαίνει εκεί και να συναντήσουμε όλους ε, που μας ενδιαφέραν, τον πρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Ορτέγα, τη σύζυγό την κυρία Μουρίγιο, επικεφαλής κοινωνικών κινημάτων, φοιτητικών, αγροτικών, εκπροσώπους με κυβερνητικών οργανώσεων, μητέρες των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στις διαπραγματεύσεις, συναντήσαμε πολιτικούς κρατωμένους, επισκεφθήκαμε τις φυλακές. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητική, καταπληκτική επίσκεψη, φορτισμένη, αλλά και πλήρης πληροφοριών. Και πραγματικά ε, την αντιμετωπίσαμε με πολύ πάθος, γιατί αυτά που συμβαίνουν εκεί είναι πολύ σοβαρά. Από τις διαδηλώσεις που έγιναν πέρυσι τον Απρίλιο, η χώρα αντιμετώπισε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μία ρήξη ουσιαστικά του δημοκρατικού συστήματος. Υπάρχει σαφής φήμωση και καταπίεση των ελευθεριών έκφρασης, συνεταιρείστε, συνέρχεστε γίνονται χωρίς δικονομικές εγγύησεις, δίκες πολιτικών ε, αντιπάλων, μαζικές ε, συλλήψεις και φυλακίσεις και το σοφρονιστικό σύστημα είναι βάναυσο, απάνθρωπο σε πολλές περιπτώσεις, εξευτελιστικό και μάλιστα γίνεται μια δίωξη των ε, ηγετών των κοινωνικών ε, κινημάτων. Ε, γίνεται εκφοβισμός και παρενόχληση των οικείων, των συγγενών των πολιτικών κρατουμένων, των διώξεις δημοσιογράφων. είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών που έφυγαν στην Κωνσταντίνα ή σε γειτονικέ χώρες αφαιρέθηκε η νομική προσωπικότητα μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης απελάθηκαν από τη χώρα ε, διεθνείς οργανισμοί από τους πιο σημαντικούς ε, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμη και η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ εκδιώχθηκε από τη χώρα. Επίσης, ε, οι πολιτικές συμφωνίες έχουν απαξιωθεί και κυρίως γιατί οι πολιτικές συμφωνίες με το καθεστώς του Ορτέγα έπληξαν το κύρος τους. Οι... Και κυρίως ε, απέναντι στις οργανώσεις που ζητούν ελευθερία και δημοκρατία. Επίσης, οι εσωτερικές διαμαρτυρίες φημώνονται. Υπάρχει μεγάλη καταστολή και καταποίηση και μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις και τα σημαντικά συλλαλητήρια καθώς και τους νεκρούς που είχαμε τους πρώτους μήνες η αντιπολίτευση αυτοεξορίστηκε πήγε στην Κωνσταντίνα. Όσοι έχουν παραμείνει στη χώρα ε, ουσιαστικά έχουν περάσει την παρανομία. Γιατί η κατάσταση αποδεικνύει μία ε, φοβερή ρήξη στην άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών. Η επισκοπική διάσκεψη, δηλαδή η Καθολική Εκκλησία, είναι πολύ σημαντικό διαμεσολαβητή και θα συνεχίσει να είναι και στο μέλλον. Η διάσκεψη των επισκόπων στην Ικαράγουα Η Επισκοπική Σύνοδος είναι απαραίτητη, ε, απαραίτητο τμήμα του διαλόγου και επίση ο νούνσιος του Βατικανού και οι επίσκοποι της Νικαράγουας παίζουν πολύ σημαντικό και απαραίτητο διαμεσολαβητικό ρόλο στην πολιτική διαδικασία της Νικαράγουας και η σημασία τους θα είναι πολύ μεγάλη και στο μέλλον. Η κυβέρνηση δείχνει μια πολύ φαλκιδευμένη εντύπωση πραγματικότητας. Η εικόνα που δίνουν είναι ότι τα Ηνωμένα Έθνη ενορχίστρωσαν ουσιαστικά ένα πραξικόπημα, ένα ιονί πραξικόπημα και το αφήγημα της κυβέρνησης είναι παρόμοιο με αυτό της Βενεζουέλας. Ουσιαστικά κατηγορούν τους Γιάνκης, όπως τους λένε, για όλα τα κακά, τα κακοσκήμενα Και αυτή είναι μια πολύ ε, παραποιημένη περιγραφή της πραγματικότητας. Και το είπα και στον πρόεδρο Ντανιέλ Ορτέγα, ότι είναι τελείως αναλυθής αυτή η εκδοχή που μας παρουσιάζει πραγματικότητα η κυβέρνηση της Νικαράγουας και οι εκθέσεις των Οργανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δείχνουν πόσο ψευδής είναι αυτή η περιγραφή της πραγματικότητας. Έχει εκραγεί η Νικαράγουα με πολλούς και διάφορους τρόπους. Φοιτητέ, αγρότες, νέοι, κοινωνικές οργανώσεις, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε μια χώρα με υψηλή πολιτική παιδεία που διεκδικεί ελευθερία, δημοκρατία και δεν αντέχει το μονοπόλιο μιας εξουσίας που έχει γίνει πια απολυταρχική ολοκληρωτική. Αυτή είναι η αλήθεια. Το τελικό συμπέρασμα της, αποστολή της αποστολής μας, για να με μακρηγορό, είναι ότι έχουμε δύο διαφορετικές Νικαράγουες που συμβαδίζουν. Υπάρχει ε, το κίνημα των Σαντινίστας, αλλά πέραν αυτού του κινήματος που έκανε την ε, επανάσταση κατά του Σωμός, έχει εγκαταλείψει τον Ντανιέλ Ορτέγα. Ο Ντανιέλ, ο Ντανιέλ Ορτέγα περιστοιχίζεται από μια ομάδα που μοιράζεται μεταξύ της ε, την ε, εξουσία με οικογενειακά και συντεχνιακά συμφέροντα και βέβαια υπάρχει αυτό το, αυτή η μνήμη και γι' αυτό της Επανάστασης και γι' αυτό ένα 20-25% των πολιτών τον στηρίζει ακόμη. Αλλά υπάρχει και η άλλη Νικαράγουα, από τους Πριτάνιους των Πανεπιστημίων μέχρι τους φοιτητές των ε, σχολών, από τους αγρότες μέχρι τα κοινωνικοπολιτικά κινήματα που διεκδικούν και απαιτούν δημοκρατία και ελευθερία. Θα πρέπει να συνεννοηθούν λοιπόν αυτά τα δύο διαφορετικά τμήματα, αυτέ οι δύο διαφορετικέ Νικαράγουε. Οπότε τα συμπεράσματά μου είναι, καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποσαφηνίσει, να αποκρυσταλώσει τη θέση της και να καταγγείλει κατηγορηματικά την ε, απολυταρχική παρεκτροπή του καθεστώτος του Ντανιέλ Ορτέγα. Και το αναφέραμε και στο ψήφισμα της 31ης Μαΐου του 2018. Θα πρέπει όμως να το επαναλάβουμε και να το διατρανώσουμε. Αποσαφηνίζοντας την πολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η καταγγελία αυτή, αυτή η καταδίκη του Ορτέγα θα πρέπει να συνοδευτεί και από επιβολή κυρώσεων προς το καθεστώς αν δεν αλλάξει. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς προειδοποίησε τον Ντανιέλ Ορτέγα ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ή θα προσφύγει στους μηχανισμούς για να πιέσει τη χώρα υπέρ της δημοκρατίας. Αλλά μόνο στα λόγια έμεινε. Και το Δεκέμβριο το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών ε, και η εκπρόσωπος Μαγκερίνη προειδοποίησε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Προειδοποίησε μόνο όμως. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Κοινοβούλιο θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσει τη θέση του και να αποκρισταλώσει μετά από αυτήν την επίσκεψη και να δείξουμε πυγμή, σθένος και να καταδικάσουμε δρυμύτατα ε, την κατάσταση αυτή ζητώντας την επιβολή κυρώσεων ε, κατά του καθεστώτος, αν δεν αλλάξει η πολιτική. Τρίτον, θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ικαράγουα να βρει το δρόμο του συμφώνου της ε, συμπεφωνημένης ειρηνικής και δημοκρατικής λύσης. Και φαντάζομαι θα ξέρετε κι εσείς, ε, οι γονείς των νεκρών παιδιών, οι σουίτε, οι Πριτάνοι των Πανεπιστημίων, οι φοιτητέ ζητούν αλήθεια και δικαιοσύνη. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις τους. Αλήθεια και δικαιοσύνη. Βέβαια η δημοκρατική διαδικασία κατά τη γνώμη μου είναι πιο σημαντική και από αυτή την άποψη η δική μας αποστολή, η κοινοβουλευτική μας αντιπροσωπεία που, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν όλες οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την ΚΟΕ μέχρι το ΕΛΚ Είχαμε ακόμη και μέλος ε, τη FDT, φιλελεύθερους ε, σοσιαλιστές. Είχαμε μια ευρεία πολιτική εκπροσώπηση και ζητήσαμε κατεπήγοντος τρία την από την κυβέρνηση. Να απελευθερώσει πολιτικούς κρατουμένους ή να μετατρέψει την προσωρινή φυλάκιση σε προσωρινή ελευθερία. Γιατί η χώρα, στη χώρα το λένε ε, οίκος έναντι φυλακής. Όσοι αναμένουν τη δίκη τους και μερικές φορές αυτές οι δίκες είναι και αβάσιμες νομικά, να βρίσκονται τουλάχιστον στο σπίτι τους και όχι στη φυλακή ενώπιον της, ενώπιση της δίκης τους και να μην ε, κακοποιούνται στη φυλακή επίσης. Επίσης ζητούμε ελευθερία διακίνησης των ε, ηγετών των κοινωνικών κινημάτων. Και τρίτον ζητήσαμε επιστροφή στην Ικαράγουα των διεθνών οργανώσεων. Αυτές είναι οι χειρονομίες ε, που θα πρέπει να ε, συνοδεύσουν τον διάλογο που θέλουμε να προωθήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περασμένη εβδομάδα πήγα και στο Μεξικό και εκεί συναντήθηκα με την ηγεσία της χώρας, γιατί και το Μεξικό είναι μια πολύ σημαντική χώρα και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Όπως κάνει και στην περίπτωση της Βενεζουέλας, θα μπορούσε και εκεί να γίνει ο διαμεσολαβητής για να βρεθεί μια συμπεφωνημένη λύση. Και εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια εμπειρογνωμοσύνη στην στον οδικό χάρτη προς τη... και στον δρόμο προς ελεύθερες εκλογές και δημοκρατικές. Να εξασφαλίσουμε τη διοργάνωση αξιόπιστων και ελεύθερων εκλογών με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, εξασφαλίζοντας ε, θεσμούς που θα μεριμνούν για την απρόσκοπτη διενέργεια τέτοιων ελεύθερων εκλογών και επίσης οι πολιτικές παρατάξεις που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία ε, συμμετέχουν στην εκπόνηση ε, ενός σχεδίου ψηφίσματος που θα υποβάλουμε στην πρώτη Ολομέλεια του Μαρτίου στο Στρασβούργο. Και στο ψήφισμα αυτό θα επιβεβαιώνουμε ουσιαστικά όλες αυτές τις ιδέες και τις συστάσεις που σας ανέφερα. Θα πρέπει να απαιτήσουμε από το καθεστώς του Ντανιέλ Ορτέγα ρεξικέλευτες αλλαγές με βάση αυτές τις τρεις προϋποθέσεις, την ελευθερία για τους πολιτικούς κρατομένους, ελευθερία διακίνησης των ε, κινημάτων και επιστροφή των διεθνών θεσμών και οργανώσεων στη χώρα. Επίσης, να διευκολύνουμε το διάλογο και αν γίνει ο διάλογος να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν γίνει να επιβάλλουμε κυρώσεις και μάλιστα αυστηρές. Αυτά είναι τα συμπεράσματα της αποστολή μα στην Ικαράγου. Ευχαριστώ. Thank you, dear Ευχαριστώ, κύριε Χαβουδέγγι. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι με τα συμπεράσματα που αναφέρατε. Ήταν μια σημαντική επίσκεψη αντιπροσωπεία για την Νικαράγουα. Έχει κάποιο κάποια σχόλια για αυτά που μα είπε ο κ. Χαουρέγγι. Όχι. Ευχαριστώ για την ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη της ειδικής αντιπροσωπείας ε, στην Νικαράγουα τον Ιανουάριο. Συνάδελφοι, έχουμε ακόμα το σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη. Ενημέρωση τώρα για την αποστολή στην Γουατεμάλα από την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τη σχέση με την Κεντρική Αμερική 29 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου. Τότε ο κ. Σταγιάν είχε ζητήσει να σταλεί αντιπροσωπεία από το Κοινοβούλιο για να εξεταστεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίω των ηθαγενών κοινοτήτων. Απουσία της κυρία Σακοράφο, ο Χαβιέ Μπενίτο, ελπίζω να, να προέφερα σωστά το όνομά σα, που επίση μετέσχε στην αντιπροσωπεία, θα μα ενημερώσει σχετικά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και της Αντικροσωπείας της Κεντρικής Αμερικής. Με χαρά θα σας παρουσιάσω τα ευρήματα της επίσκεψης της αντιπροσωπείας στη Γουατεμάλα μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2018. Αντιπροσωπεία που όπως είπε ο Πρόεδρος είχε σαφ, τρεις στόχου στόχους. Πρώτον εξέταση της κατάστασης ε, με την ε, της ε, Επιτροπής Αλήθειας και την απόφαση του Πρόεδρου τότε να μην ανανεώσει την εντολή του ΟΗΕ για την Επιτροπή Ατιμωρησίας, κατά της Ατιμωρησίας, την εξέταση της διαδικασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως εις βάρος των υπεραστηρικτών των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τρίτον, οικονομικά και πολιτικά θέματα με την χώρα αυτή και την Κεντρική Αμερική ευρύτερα. Πρώτον, γενικά συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η κυβέρνηση είναι πολύ κλειστή με την οποία η διπλωματική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων είναι πολύ σύνθετη. Μιλήσαμε με κυβερνητικούς εκπροσώπους, και υπουργούς, οι οποίοι μιλούσαν συνεχώς, αναφέρονταν συνεχώς στην εθνική κυριαρχία και φάνηκε ότι η δουλειά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα συνεργασίας στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου αντιμετωπίζεται ως επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. Τούτο περιγράφει ε, εν πρώτης μια σύνθετη διπλωματική σχέση με την κυβέρνηση της χώρας. Σε ένα πλαίσιο πολιτικό και κοινωνικό σύνθετο. Πολιτικά, λόγω της ε, καμπής, ε, της αλλαγής της, της θέσης της κυβέρνησης, που ενώ προεκλογικά υποστήριζε το ΣΥΣΙΚ, την ε, Διεθνή Επιτροπή κατά της Ατιμορρησίας, σε μια συνέντευξη τύπου του Προέδρου, παρουσία και στρατιωτικών απέριψε την επιτροπή αυτή. Ταυτόχρονα η χώρα έχει υψηλότατα επίπεδα και ε, υποσυτισμού και εγκληματικότητα. Είναι βέβαιο ότι η Γουατεμάλα έχει σημαντική ανάπτυξη, 3% το χρόνο περίπου, αλλά συνεχίζει μια τεράστια ανισότητα και εξαιρετικά χαμηλή φορολογήσει ε, από τις χαμηλότερες στην Κεντρική Αμερική. Κάτι που δεν μπορεί να εξασφαλίσει υποστήριξη από το δημόσιο στην αντιμετώπιση της ανισότητας που αφορά κυρίως τους αυτόχθονες λαούς της Γουατεμάλας. Για να μπούμε λίγο περισσότερο στα θέματα της Επιτροπής κατά της Ατιμορρησίας, του ΘΙΣΙΓ. Το 2017 η φύση ήταν, ε, είχε κομβικό ρόλο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Ε, η εισαγγελική αρχή αυτή έφερε στην ε, παρέπεψη δικαιοσύνη περίπου 300 περιπτώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων, πρώην πρόεδρος της Γονεμάλα μεταξύ των οποίων, ο οποίος τώρα είναι ο πρόεδρος, αλλά και τον τωρινό πρόεδρο κ. Μοράλες. Συνεχίζει να λειτουργεί χάρη στη διεθνή χρηματοδότηση που κατά βάση προέρχεται από δύο φορείς, δύο πλευρές της ΕΠΑ που πάντα υποστήριξαν το ΣΥΣΙΓ ακόμα και επί προεδρίας Τραμπ παρότι μειώθηκε κάπως και ακόμα περισσότερο από μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 166 εκατομμύρια δώσαμε στην ΣΥΣΙΓ η συνεργασία του κράτους με το ΣΥΣΙΚ διακόπηκε σε τρεις βασικές στιγμές. Πρώτον, αναγγελία της μη παράταση της εντολής ε, της Επιτροπής ε, τον Αύγουστο, απέλαση του κ. Βελάσκες από τη χώρα που κρίθηκε ως ε, persona non grata και μονομερή διακήρυξη τον Ιανουάριο του 18, το Δεκέμβριο του 18 της διακοπής της συνεργασίας με τη ΦΥΣΙΚ. Εμείς τονίσαμε, ε, υπογραμμίσαμε ότι η προεκλογικά ο κ. Μοράλες ήταν υπέρ του ε, κάτι που άλλαξε όταν ε, η εισαγγελία απήγγελε κατηγορίες εναντίον ε, του ίδιου, του αδελφού του και του γιού του για διαφθορά. Από τότε ξεκίνησε ε, μια καμπάνια κατά του ΘΥΣΙΚ ενώ διώχθηκαν από την κυβέρνηση υπουργοί που ήταν υποστηρικτές της. η, η Ένωση και η διεθνής κοινότητα για να βοηθήσουν την μάχη κατά της ατιμοδησίας ε, και της διαφθοράς πρέπει να επιμείνουν ιδίω ε, σε κάποιες περιπτώσεις και με λιγότερο διπλωματικούς τρόπους ασκώντας μεγαλύτερη πίεση σε κάποιους εκπροσώπους της Γουατεμάλας. Ανθρώπινα δικαιώματα ιδίως τις συγκρούσεις για την ιδιοκτησία της γης και την ε, δολοφονία ή παραπομπή σε δίκη υποστηρικτών ε, των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη Γουατεμάλα. Το 60% του πληθυσμού είναι αυτόχθονες, αλλά δεν μετέχουν στην πράξη στην πολιτική διαδικασία, είναι αποκλεισμένοι και εξαιρετικά φτωχοί στη μεγάλη πλειοψηφία τους. Οι δηλώσεις του Πρόεδρου την Άνοιξη του 18 ε, όταν χαρακτήρισε πολλές οργανώσεις αυτοχθόνων ως τρομοκρατικές, οδήγησαν σε αύξηση της βίας. Και από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 όταν πήγαμε εκεί, 24 ηγέτες, το αυτόχθονοι ηγέτες, δολοφονήθηκαν. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εγκληματίες δεν συνελήφθησαν. Αυτό το τονίσαμε πολλές φορές, αλλά η, και ο πρόεδρος και οι υπουργοί κάνουν το ίδιο πράγμα. Θεωρούν ότι αυτές οι πολιτικές δολοφονίες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της εγκληματικότητας στην, της γενικότερης εγκληματικότητας στη χώρα, αγνοώντας την πολιτική διάσταση των φόνων αυτών. Αυτό το είπαν, το έλεγαν όλοι, με τρόπο έως και προσβλητικό σε κάποιες περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά τους, οι οργανώσεις των αυτοχθόνων ε, ζήτησαν τα εξή Πρώτον, δικαίωμα ε, διαβούλευσης όπως περιγράφεται στην σύμβαση του 79 του ε, Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που έχει επικυρώσει η Γουατεμάλα και δεύτερον μηχανισμούς ελέγχου της λειτουργίας των πολυεθνικών, των ευρωπαϊκών πολυεθνικών στην ευθύνη των συγκρούσεων. Ξέρετε πολλές συγκρούσεις έχουν να κάνουν με την κατανομή της ιδιοκτησίας της γης. Το 10% του πληθυσμού έχει 80% της ιδιοκτησίας της γης στην Γουατεμάλα. Τούτο οφείλεται εν πολλής στον τρόπο με τον οποίο δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη οι συμφωνίες ειρήνης του 1996. Τονιζόταν Ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε το δεχόμενο κυρώσεων προς τη, κυβέρνηση της Γουατεμάλας στο πλαίσιο αυτό. Η διεθνής κοινότητα ε, συνεργάζεται με την ομάδα C3 που, C13 ε, συγγνώμη, που παρακολουθεί τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου με παρακολούθηση ειδικών, ε, το, επιτόπιες επισκέψεις. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντική, όπως και η ομάδα Φίλτρο. Οι δύο αυτές οργανώσεις κάνουν πολύ καλή δουλειά και νομίζω η επίσκεψη της Ένωσης βοήθησε το έργο αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να υποστηρίξουν ακόμη περισσότερο η Ευρώπη. Λολίτα Τσάβες τώρα, το βραβείο Ζαχάροφ, ε, η φιναλίστος στο βραβείο, στο βραβείο Ζαχάροφ, δεν είναι δυνατή η ασφαλής επιστροφή της, ε, επιστροφής της ε, στην Γουατεμάλα και κανείς από την κυβέρνηση δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον <coughs> για την προσωπικότητα αυτή που αναγνώρισε και το Κοινοβούλιο και ο πρόεδρος κ. Σταγιάννη. Τελευταίο θέμα, συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Γουατεμάλα. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε δύο έργα που χρηματοδότησε η Ένωση, εξοπλισμός μιας φυλακής γυναικών ε, και ανηλίκων και δεύτερον πρόγραμμα ε, επαγγελματική κατάρτισης. Η συνεργασία αυτή προφανώ δεν μπορεί να λύσει τα βαθιά ριζωμένα προβλήματα της ανισότητας στη χώρα, αλλά διαπιστώσαμε ότι η συνεργασία αυτή βελτιώνει την σημερινή κατάσταση κάποιων ομάδων, κάποιων συγκεκριμένων περιπτώσεων ή κομματιών του πληθυσμού η Ένωση κάνει καλή δουλειά στον τομέα αυτό και θεωρούμε σημαντικό να συνεχίσουμε την υποστήριξη στο έργο αυτό. Προς το παρόν η Γουατεμάλα είναι η δεύτερη χώρα σε ε, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θετικό όπως σας είπα αυτό, διαπιστώνουμε ωστόσο ότι η συνεργασία με την κυβέρνηση της χώρας είναι κάτι πολύ περίπλοκο ακόμα και σε πολύ συγκεκριμένα απλά χαρακτηριστικά της συνεργασίας αυτής. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια και έλλειψη ενδιαφέροντος σε μεγάλο βαθμό των εθνικών αρχών για τη συνεργασία αυτή. Υπάρχουν προβλήματα σε απλά πράγματα. Πώς εισάγεται σε ένα λιμάνι ε, της Γουατεμάλας υλικό για να χρησιμοποιηθεί στην φυλακή που επισκεφθήκαμε η συνεργασία επέτρεψε να μηχανογραφηθεί όλη η ενημέρωση για τα στοιχεία για τους φυλακισμένους πριν τα στοιχεία αυτά ήταν σε, μια, σε ένα γραφείο, το ένα έγγραφα πάνω στο άλλο. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ολοκληρώσει την ποινή του, αλλά κανεί δεν το ήξερε και παρέμειναν μέσα. Υπήρχαν τέτοια προβλήματα και γραφειοκρατικά εμπόδια που σε συνδυασμό με την αδιαφορία που προανέφερα δημιουργούν προσκόμματα στην συνεργασία. 80 εκατομμύρια ευρώ που, είχαν, που έχουν χορηγηθεί για τη μετώπιση του υποσυτισμού δεν αναλώθηκαν. Τελειώνω. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη συνεργασία με τη Γουατεμάλα. Πιστεύουμε ότι οι ομάδες των χωρών στην ομάδα φίλτρο ε, κάνουν καλή δουλειά στην προσπάθεια παρακολούθησης ε, και προστασίας των δικαιωμάτων ανθρώπου και των υπερασπιστών του. ωστόσο βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα όπως η Επιτροπή κατά της Εντιμοδησίας που πρέπει να μας απασχολήσουν ε, και να μας οδηγήσουν σε μια πιο στιβαρή διπλωματική στάση έναντι της κυβερνήσεως της χώρας από πλευράς της διεθνούς κοινότητας. Κλείνω ευχαριστώντας όλη την ομάδα της γραμματείας που κατέστησε δυνατή την επίσκεψη αυτή. Τον Φρέντερικ για παράδειγμα που μας βοήθησαν ε, στην ε, επίσκεψη και τον ε, πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριο Στέφανο Γκάτο, για την πολύ καλή δουλειά και εξαιρετική υποδοχή που μας προσέφερε. Δεν είναι εύκολη δουλειά να είσαι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γουατεμάλα. Οι σχέσεις, οι διπλωματικές σχέσεις των δύο πλευρών είναι πολύ σύνθετες όπως σας είπα και αυτός κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ αγαπητέ για την παρουσίαση αυτή των πεπραγμένων ε, της επισκεψής σας στη Γουατεμάλα. Πολύ ενδιαφέρουσα η αντίληψή σου για το πώς έχει κατάσταση στη χώρα και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω όποιον συνάδελφο ενδεχομένω θέλει το λόγο για να διατυπώσει σχόλια παρατηρήσεις. Ο κ. Χαουρέγγι, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση έχω. Προβλέπετε στο πλαίσιο της ΔΕΚΑΜ να κατατεθεί στην Ολομέλεια μια πρόταση να κάνουμε μια ε, χειρονομία εμείς ως κοινοβούλιο, ίσως στην Ολομέλεια, δεν ξέρω, ίσως ε, μέσω της διαδικασίας ε, του κατεπήγοντος, της συζήτησης των επιγόντων ή με συζήτηση και ψήφισμα. Γιατί πραγματικά το ότι ε, πλέον δεν μπορεί να είναι εκεί ότι εκδιώχθηκε η θήθη η Επιτροπή για τα φαινόμενα τιμωρησίας και το ότι δεν μπορεί να παρατηρεί τα φαινόμενα επιτόπου είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν προβλέπεται και αν δεν προβλέπεται θα ήθελα να το θέσω ως ιδέα να γίνει μια σύντηση. Ο κύριος Μπενίτο πράγματι μας απασχόλησε ως αντιπροσωπεία μεταξύ άλλων το να προωθήσουμε ίσως την κατάθεση ενό ψηφίσματος από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω το 2017 ήταν που είχε κατατεθεί ένα ψήφισμα κατεπίγοντος για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα. Εκεί πολλοί φορείς μας εξέθεσαν τη σπουδότητα του ψηφίσματος αυτού και συμφωνούσαν και αυτοί ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένα δεύτερο ψήφισμα κατεπήγοντος. Συμφωνώ και εγώ, είτε κατεπήγον, είτε ψήφισμα και συζήτηση. Ιδίω ε, για την ε, εκδίωξη της ΣΥΣΙΓ, ε, της Επιτροπής κατά της Ατιμορφίας. Επιτροπός Μογκερίνη έχει προβεί σε μια ανακοίνωση ήδη. Καλό θα ήταν και σκόπιμο να ακολουθήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα αντίστοιχο διάβημα. Βέβαια, σε αυτή τη δήλωση ε, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι έχουμε προεδρικέ εκλογέ στη Γουατεμάλα τον Ιούνιο, άρα δεν υπάρχει πολύ χρόνο και θα πρέπει τάχιστα το Κοινοβούλιο, αν είναι, να καταθέσει αυτό το ψήφισμα. Και με τον κίνδυνο να ειδωθεί αυτό ως παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας. Η Γουατεμάλα περιλαμβάνεται στο φετινό κατάλογο πιθανών χωρών στις οποίες ε, θα μεταβεί η Επιτροπή Εκλογικής Παρατήρησης. Βέβαια πρέπει να μας καλέσει η κυβέρνηση και με την εμπειρία που αποκόμισα δεν το βλέπω και τόσο πιθανό κάτι τέτοιο. Αλλά θεωρώ ότι μια Επιτροπή Εκλογικής Παρατήρησης εν της πόλωσης ε, της βίας ε, πρώτων εκλογών και η θέση ίσως και των όπλων δυνάμεων στην κυβέρνηση και της ε, ισχύω που αποκτούν είναι ένα θέμα. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ο πρόεδρος, ωραία. Σας ευχαριστώ. Βλέπω ότι συνεχίζετε το μεταξύ σας διάλογο. Φυσικά το ζήτημα της ε, Γουατεμάλα και της Κεντρικής Αμερικής εν είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί στην Ολομέλεια. Είναι θέμα των ε, πολιτικών ομάδων να αποφασίσουν κατά πόσο μπορούμε να έχουμε συζήτηση ή όχι. Σας ευχαριστώ πάντως ε, για τις πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις και τις δύο. Δεν έχω κάποιο αίτημα. Να σας πω λοιπόν ότι θα συνεχιστεί απόψε το μεσημέρι στις 3 ώρα η συνεδρίασή μας με μια μακρά ε, σειρά ψηφοφοριών. Ε, πάντως η πρωινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο. Καλό μεσημεριανό διάλειμμα λοιπόν.